Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην ε, ψηφοφορία για να μπορέσουμε να φάμε σχετικά νωρί. Το επόμενο σημείο είναι η ψηφοφορία βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας, ε, η πρώτη από τις πέντε εκθέσεις για την έκθεση της κυρίας Ματέρα, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. να καθίσει. Ένα λεπτό. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η επόμενη έκθεση της κυρίας Ματέρα για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής ε, στην παγκοσμιοποίηση. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας εγκρίθηκε. Πάλι μια έκθεση της κυρίας Ματέρα, πάλι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 43 από την Ιρλανδία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία εγκρίθηκε και τελευταία έκθεση της κυρίας Ματέρα για το ίδιο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αίτηση EGF 2011, 80 Lower από την Άνω Αυστρία. Παρακαλώ ψηφίστε, ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε Έχω παραλείψει μια έκθεση, συγγνώμη, αλλά γύρισα πολύ γρήγορα τη σελίδα. Ξεχάσαμε την Ελλάδα. Ελλάς. Ε, παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κυρία Ματέρα. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό την Ελλάδα. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του κυρίου Κασμαρέκ για την ε, Μεκτή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και 2010 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην έκθεση της κυρίας Παλιαδέλη για το Ευρωπαϊκό Σήμα Κληρονομιάς. Τροπολογία 1, ονομαστική ψηφοφορία, της ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Άρα εγκρίνεται η θέση του Συμβουλίου. Συγχαρητήρια κυρία Παλιαδέλη. Περνούμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Σερακιάνη για την ενιαία, στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο. Μου ψηφοφορεί για όλες τις τροπολογίες της Επιτροπής Μεταφορών. Παρακαλώ, ψηφίστε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται, 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Ε, επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 51 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση 52, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 54 κατά τμήμα η ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Με ονομαστική ψηφοφορία το δεύτερο τμήμα. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίθηκε. Η 67 σε δύο τμήματα. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της 67. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Ε, ε, ε, ευρύτατη πλειοψηφία υπέρ. Δεύτερο τμήμα τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. εγκρίνεται. 98 σε τρία τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση 151. Επαλήθευση παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Απερίφθη με συντριπτική πλειοψηφία. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Είναι όλες με ονομαστική ψηφοφορία. 136 πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρας. Δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Άρα καταπίπτει το τρίτο τμήμα. Και περνάμε στην τροπολογία 53 που έχουμε και προφορική τροπολογία του κυρίου του... Τρεμόζα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Πού είναι ο κύριος Τρεμόζα. Doesn't go. It does. Yes. Thank you. Λειτουργεί. Ωραία. Ευχαριστώ. Είμαι ο Σκιώδης των Φιλελευθέρων για αυτή την έκθεση. Οι Φιλελεύθεροι θα ήθελαν να καταθέσουν μια προφορική τροπολογία στην τελευταία ε, ε αράδα του άρθρου. Θέλουμε να βελτιώσουμε το κείμενο προσθέτοντας τέσσερις μονολέξεις. Μετά το capital employed μπορούμε να προσθέσουμε εκτός από ότι είναι δημόσια χρηματοδότηση, except from public funding. Και νομίζω ότι οι σκιώδεις εισηγητές των λοιπόν πολιτικών ομάδων συμφωνούν. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος, υπάρχουν ενστάσεις ε, ως προς την προφορική τροπολογία. Να δούμε πόσοι βουλευτές ε, έχουν ε, εγερθεί. Έχουμε 40 νομίζω. Άρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 53 τώρα σε τρία τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρα το πρώτο τμήμα, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης. 137 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 Επαλήθευση εφόνο, ε, για την 137 εφόσον το ζητάτε. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Καταψήφισαν οι φιλελεύθεροι. Αυτό έπρεπε να κάνουμε μάλλον. 153 υπέρ κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 62 και 162 μαζί για την ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συγγνώμη, υπάρχει ένα αντίστοιχο τμήμα, έτσι μου λένε, το λένε, δεν ξέρω τι είναι, υπέρ κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Αυτά είναι τα αντίστοιχα τμήματα της 162 τώρα. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τώρα στο αντίστοιχο τμήμα της 62. Ψηφίζουμε επαλήθευση. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Αυτό είναι χειρότερο για τους πίνακες που έχουν ε, όταν είναι να πάρει κανείς το τρένο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ε, αντίστοιχο τμήμα της 162 τώρα, παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, το αντίστοιχο τμήμα της 62, σε δύο τμήματα κιόλας. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 62 και 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Για φαντάσου. Ξανά. Ξανά λοιπόν τα αντίστοιχα τμήματα της 62 και 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι εγκρίνονται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Για την 141 παρακαλώ ψηφίζετε. Πέρας. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 159 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Δεν είναι σωστό. Συγγνώμη. 159 υπέρ, παρακαλώ, το κάνουμε πάλι. Κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συγγνώμη. ζωαβή ε, μου θυμίζει αυτό. Να ελέγξουμε το αντίστοιχο τμήμα της 79. Ε, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 79. Πέρας της κοινωνικής ψηφοφορίας. Σαφής πλειοψηφία. Ψηφίζουμε τώρα το αντίστοιχο τμήμα της 79 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Α, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 163. Αρχίζει. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 142 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείται. 144 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα βάζω την πρόταση της α, Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ε, σε ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Και τώρα, το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος το θέτω σε ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχής ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Υιοθετείτε. 526 υπέρ, 80 κατά. Μπράβο κύριε Σερακιάνη. Πάμε στο ψήφισμα Durban τώρα, για τον Durban δηλαδή. Την παράγραφο 3 ψηφίζουμε σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Υιοθετείτε. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφο 8. Σε δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Αρχής ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Παραμένει ανοιχτή. Πέρας τώρα. Τη ψηφοφορία Υιοθετείτε. Παράγραφος 9. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Υιοθετείτε. Τροπολογία 9. Με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Πέρα ψηφοφορία Απορρίπτεται. Παράγραφος 10 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Παράγραφος 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 16 ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Υιοθετείται. Παράγραφος 17. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τώρα. Τροπολογία 1 και 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και οι δύο. Παράγραφος 21. Υπέρ. Κατά αποχέ. Υιοθετείτε. Πράγμα 22. Σε δύο τμήματα και με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ξεκινάει η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. ε, αρχίζει. Τελειώνει. Υιοθετείτε. Παράγραφος 23. Υπέρ. Κατά. Να το αλλάξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα γιατί δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Παράγραφος 25 σε δύο τμήματα και με ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική ψηφοφορία τώρα ξεκινάει. Πέραστη. Υιοθετείτε. 35. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Την 35. το δεύτερο τμήμα της 35. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Παράγραφος 38 με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 39. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφο 46, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, Κατά. εποχές Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. εποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 51. Παράγραφο 51. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 13. Υπέρ. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. εποχές. Απορρίπτεται. τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 64. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Το δεύτερο βήμα τη 64. Αρχής ψηφοφορία. Πέρα. Υιοθετείτε. 14 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Και τώρα το εκτιμώντα 6 ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχής ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Αιτιολογική σκέψη D, δέλτα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, υιοθετείτε. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, υιοθετείτε. Αιτιολογική σκέψη 1, σε δύο τμήματα. Όχι, όχι, συγγνώμη, δεν είναι ένα. <laughs> Ήταν I. Θέλετε να ελέγξετε το δεύτερο τμήμα του D, του D, του δέλτα. Ναι, το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Υιοθετήθηκε. Πάμε στο I σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. J, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 7, τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 7. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Διολογική σκέψη π. Σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, υιοθετείτε. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Q, υπέρ, κατά, Εποχές, διοθετείτε. Και τώρα θέτω το τροποποιημένο ψήφισμα σε ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει. Πέρας. διοθετείτε, Με τεράστια πλειοψηφία. Και τώρα πάμε στη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Πάραφο 3 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. <laughs> Δεν υπάρχει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ε, το άλλο το εφηβρέγω. Πάραχος A. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. Παράγραφος 12. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Και τώρα βάζω το ψήφισμα ε, σε ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Σχεδόν τελειώσαμε. Σχεδόν. το επόμενο σημείο είναι η έκθεση Μπόρις για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή. Πριν ψηφίσουμε όμως, θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μπόρις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου εδώ. Και αυτή η έκθεση έρχεται να συμπληρώσει το βραβείο Λουξ. Σε μια εποχή κρίσης είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι ε, προς τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Η βιομηχανία του κινηματογράφου στην Ευρώπη περιμένει εδώ και 10 χρόνια αυτή την έκθεση. Και αν την υιοθετήσουμε, θα επιταχύνουμε τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και οι Ευρωπαίοι θα έχουν καλύτερη πρόσβαση ε, στο κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους θα ψηφίσετε υπέρ. Ευχαριστώ. Παράγραφος 9, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 17. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 21. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Πού έχω φτάσει. 35 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 36 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 69 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε Δεύτερο τμήμα προ, υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 92 με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει τώρα. Πέρας της. Υιοθετείτε. 93. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 119. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Ομοφωνία. 123. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 125. Υπέρ κατά εποχές υιοθετείται. Θέτω το ψήφισμα σε ψηφοφορία. Με η ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρας της ψηφοφορία Υιοθετείτε μια τεράστια πλειοψηφία. Μπράβο κύριε Μπόρις και μπράβο στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο.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 Okay, we're coming to explanations of vote now. Θα έρθουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. On the Katsmarek report. Κυρία Σιλβέστρης. Την έκθεση Κατσμάρεκ.